Allora, buongiorno. Χαίρετε. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι και επαναλαμβάνετε η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία διεκόπη στις 4 Ιουλίου του 2019. Να καλωσορίσω και το κοινό το οποίο είναι εδώ στα θεωρία για να παρακολουθεί την έναρξη της Ολομέλειας στα πρακτικά τα έγγραφα τα οποία εγκρίθηκαν ε, στις 4 Ιουλίου του 2019 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν ε, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Κάποιες ανακοινώσεις τώρα. Μετά από την εκλογή του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι χειρεύει η θέση του από τις 7 Ιουλίου του 2019. Οι αρμόδια αρχές των κάτω χωρών μου διαβίβασαν την εκλογή της κυρίας Λάρα Βόλτερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα αντικαταστήσει τον κύριο Φρανς Τίμερμανς, από τις 4 Ιουλίου του 2019. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδος μου ανακοίνωσαν την εκλογή του κυρίου Εμμανουήλ Φράγκου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αντικαθιστά τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο από τις 10 Ιουλίου του 2019 να καλωσορίσω τους νέους συναδέλφους και να υπενθυμίσω ότι ε, απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανα του, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό μας. Έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα και από το ECR κάποια αιτήματα τροποποίησης ε, της σύνθεσης των επιτροπών ονόματα θα βρίσκονται στα πρακτικά της ε, παρούσας ε, συνεδρίασης. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι ορισμοί αυτοί θεωρούνται εγκεκριμένοι. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Κόρμπετ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε τα ονόματα κάποιων μελών που έχουν ήδη αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο. Είστε βέβαιος ότι εκεί δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί το σύνολο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που από ό,τι φαίνεται απουσιάζει. Ε, πολύ λεπτό το χιούμορ σας. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Το οριστικό σχέδιο ημερήσια διάταξη, το οποίο εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στι 11 Ιουλίου βάσει του άρθρου 157, σα έχει διανεμηθεί. Για την Τρίτη, αύριο δηλαδή, η ομάδα της GUNGL έχει ζητήσει η δήλωση τη υπάρξη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι Εξωτερικέ Υποθέσει και την Πολιτική Ασφαλεία για την κατάσταση στη Βενεζουέλα να μην ολοκληρωθεί με ψήφισμα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βίλα Ναβαρούιθ για να παρουσιάσει το αίτημα εξ ονόματο τη ομάδα σα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, εξ ονόματος Ενωτική Αριστερά, ζητούμε να αφαιρεθεί το ψήφισμα από την ημερήσια διάταξη για τη Βενεζουέλα. Η συζήτηση να παραμείνει, βεβαίω το θεωρούμε απαραίτητο, αλλά αυτή τη στιγμή που ζούμε με μια νέα διαδικασία διαλόγου που έχει προωθήσει η Νορβηγία και όπου εμπλέκονται όλοι οι φορεί και προχωρούν οι διαπραγματεύσει. Μέχρι και ο ίδιο ο Πάπα τι έχει στηρίξει. Είναι ευκαιρία λοιπόν για το Κοινοβούλιο να σταματήσει να βγάζει ψηφίσματα και να προσπαθεί να αναμειγνύεται στα εσωτερικά της Βενεζουέλας και να ε, φανεί πρωταγωνιστή στην υπεράσπιση του διαλόγου, της ειρήνης για να μπορέσει να βοηθήσει χωρίς καμιά αμφιβολία με τη μόνη οδό για να υπάρξει μια κατάσταση μόνιμη υπέρ του λαού της Βενεζουέλας. Ευχαριστούμε κυρία Βιλανουεβα Ρουιθ. Να δώσω το λόγο σε κάποιον ο οποίος ε, θέλει να παρέμβει για να εκφράσει την αντίθεσή του. Ο κύριος Γκάλερ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα να απορρίψουμε αυτό το αίτημα. Βεβαίως και μπορούμε στο ψήφισμά μας να σημειώσουμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ε, για ότι υπάρχουν και πρωτοβουλίες τις οποίες και να καλωσορίσουμε. Αλλά πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι δραματική και είναι σαφές ότι είναι δραματική. Οπότε μπορούμε να ε, ε, εκφράσουμε άποψη και να αποφανθούμε και σε ψήφισμα. Γνωρίζουμε την τραγωδία που επικρατεί εκεί. Εκατομμύρια προσφύγων έχουν αποχωρήσει από τη χώρα και αποσταθεροποιούν τώρα και τη γειτονία ολόκληρη. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να λάβουμε θέση για την κατάσταση εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Επομένως ε, ψηφίζουμε το αίτημα της ομάδος της ΓΟΕ με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Hanno votato Ψήφισαν όλοι. Hanno votato Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Το αίτημα απορρίπτεται. Επομένως, η ημερήσια διάταξη παραμένει ω. έχει. Για την Τετάρτη τώρα, η ομάδα Γκουεντζιέλ έχει ζητήσει οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ να προσθεθούν ως ε, τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την Τετάρτη το απόγευμα μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, περιοχές ε, καθαρού αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βιλανού Ρουίφ για να παρουσιάσει το αίτημα εξ ονόματος της ομάδος της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι θεωρούμε σημαντικό να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης ε, η συμφωνία με το Μερκοσούρ που μέχρι τώρα το διαπραγματευόμαστε με όρους αδιαφανείς εδώ και 20 χρόνια. Σίγουρα θα επιδράσει ε, σε πολλές χώρες, σε πάνω από 33.000 αγρότες ε, που θα υποστούν τις νέες σκληρές συνέπειες αυτής της εμπορικής συμφωνίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει εδώ η συζήτηση την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο. Χάνσεν για την ε, αντίθετη παρέμβαση. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είμαι αντίθετος η προσθήκη αυτή στην ημερήσια διάταξη. Τα έγγραφα τώρα μόλις δημοσιεύονται, θα πρέπει να τα αναλύσουμε προσεκτικά. Η Επίτροπος Μάλστρομ ανακοίνωσε ότι θα έρθει την άλλη εβδομάδα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ΙΝΤΑ, οπότε ε, θα θέλαμε να απορριφθεί αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν το αίτημα. Διανατάσσεως χειρός. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματο της ΓΚΟΕ. Σηκώστε τα χέρια σας. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Οριστικοποιείται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Δεν υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο. Στην ημερήσια διάταξη τώρα στη συνέχεια έχουμε τις παρεμβάσεις ενός λεπτού βάσει του άρθρου 162 του κανονισμού. 172, ε, συγγνώμη. Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 184α ως πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας θα ήθελα να τονίσω ότι ο Ρόμπερ Ρόλαντ, Βρετανός Ευρωβουλευτής, την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε ένα σχόλιο που λέει ότι εν ώψη του Brexit θα πρέπει να έχει την τύχη του Μπελγκράνου οποιοδήποτε αλλιευτικό σκάφος στα ύδατα ε, της Βρετανίας. Ξέρετε ότι το 1982 στην ένοπλη σύραξη το αργεντινό αυτό σκάφος βυθίστηκε και είχε 300 νεκρούς. Πραγματικά ε, αυτό ε, το καταγγέλουμε. Και όσο απεχθεί και να είναι αυτά, υπονοούν ότι μπορούν να φωνευθούν Ευρωπαίοι αλληλείς σε ύδατα τα οποία ε, εδώ και χρόνια εκμεταλλεύονται. Η ιστορία της Ευρώπης, κύριε Πρόεδρε, δείχνει ότι έχουν νόημα και τα λόγια. Τα λόγια μπορούν να προωθήσουν την ε, φιλία, αλλά μπορούν να σφυριλατήσουν και το μίσος και το διχασμό. Πρόεδρε, ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς ε, με τη δική μου απέχθεια πραγματικά και την απόρριψη των όσων υπόθηκαν. Ευχαριστούμε κύριε Ντέιβις. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας. Ρόλαντ. Ρόλαντ. Ο κύριος Ρόλαντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που με επιτρέπετε να μιλήσω. Για να απαντήσω στον άλλο Ευρωβουλευτή θέλω να πω το εξή. Απαντούσα σε μια λεκτική επίθεση που απευθύνατε σε ένα συνάδελφό μου, σε μια συνάδελφό μου, τη Τζον Μάρμερη, όταν σας βρήκε και σας μίλησε έξω από την Επιτροπή Αλληλείας, που είστε πρόεδρος. Ε, την ε, υβρίσατε και θέλω να ε, δεχτείτε επίπληξη πειθαρχική. Αυτό απάντησα υπερασπιζόμενος τον αλλιευτικό κλάδο της Βρετανίας που συστηματικά καταστρέφεται από την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρική αλία. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υποστηρίξω και να υπερασπιστώ τους Βρετανούς ε, Πραγματικά μου ξέφυγε αυτό γιατί έχει αποδεκατιστεί η αλία μας δεν θα πρέπει να το πάρετε τη μετρητή. Φυσικά εγώ δεν είμαι υπέρ τη βία στα πελάγη, παρόλο που το είδαμε αυτό να συμβαίνει το 2018, όταν συνεπλάκησαν ε, Άγγλοι με Γάλλους αλληλεί μέσω πέλαγα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι η Βρετανία αλληλείς θα πρέπει να ε, ασκήσουν τέτοιες μεθόδους ε, εισβολής και επιδρομής σε αλληλευτικά σκάφη. Και εγώ πάντα θα τους υπερασπίζομαι. Fox. Yes. Η κυρία Ένα πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε για τη Βρετανική αντιπροσωπεία είναι ότι δεν έχουμε χιούμορ και έχει σημασία ο ελεύθερος λόγος. Είναι εξωφρενικό ότι ε, χρησιμοποιείται αυτό, αυτή η Βουλή από κάποιους ε, από το Ηνωμένο Βασάλειο για αυτά τα σχόλια, ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα πρέπει να, με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Είμαι υπέρ ε, του, της ε, ελευθερίας του λόγου του καθενός. Είναι σημαντικό και η ελευθερία είναι σημαντική και εμείς στο κόμμα του Brexit εσείς μάλλον θα, πρέπει να σημειώσετε όταν λέμε ότι εμείς θα σας περαψηφίσουμε και θα πρέπει να σταματήσετε να ε, μας ε, ενοχλείτε. Αυτό, αυτή η Βουλή δεν είναι δημοκρατική. Έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από μικροκαυγάδες ε, που ξεκινούν από τους φιλελεύθερους ενάντια στους Βρετανούς συναδέλφους. Thank you, colleagues. And on the matter Ευχαριστώ. Στο θέμα της ελευθερίας του λόγου ξεκινάμε με τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με τον κανονισμό 172 και έχω έναν κατάλογο με ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής ο κύριος Βιντσέντζε για ένα λεπτό. Ε, πρόεδρε, συνάδελφοι, στα κράτη τη μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί και νόμοι που ισχύουν ε, για την προστασία ε, των εθνικών μειονοτήτων. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ ε, δυνατές οι διασφαλίσεις, αλλού είναι κάποιο εν μέρη λύσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται καν οι εθνικές μειονότητες. Στη χώρα μου, στη Ρουμανία, ο νέος νόμος, η τροποποίηση του νόμου έχει περιορίσει ε, τις ε, διασφαλίσεις. Οι, οι κανονισμοί για την ουγγρική γλώσσα δεν υλοποιούνται. Ε, περιορίζεται η χρήση της ουγγρικής γλώσσας και είναι πολύ ανησυχητικό γιατί δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος ανάμεσα στην ρουμανική πλειοψηφία και την ουγγρική μειονότητα στη χώρα. Και εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσουμε την συνεργασία, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να υπάρχει το κράτος δικαίου για να τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί. 50 εκατομμύρια ε, μειονότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ελπίζουν ότι θα τηρούνται αυτά τα πρότυπα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κύριος Χάουαρτ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το, η ψήφος είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη στους πολίτες για να ψηφίζουν. Πριν από έξι εβδομάδες συνέβη το αντίθετο στο Ηνωμένο ε, στις η προσέλευση στις ευρωεκλογές αυξήθηκε ενώ πολλοί πολίτες που ζούσαν σε χώρες ε, όχι στις δικές τους χώρες ε, δεν κατάφεραν να ψηφίσουν. Δυστυχώς η ανταπόκριση του Ηνωμένου Βασίλειου στην κριτική ήταν αρνητική. Άρα οι αλλαγές απαιτούνται να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να απλουστευτεί η διαδικασία και να γίνει πιο εύκολη για κάθε Ευρωπαίο πολίτη να μπορεί να ψηφίζει όπου και να ζει απλά υπογράφοντας ε, μία δήλωση ε, στα κέντρα ψηφοφορίας. Ε, ζήτησα να επανεξεταστεί αυτό το θέμα πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, έτσι ώστε να έχει κάθε πολίτη το δικαίωμα να ψηφίσει όπου και να ζει. Ευχαριστώ. κυρία Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο για πρώτη φορά και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να τονίσω ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή. Τα πάντα φυσικά εξαρτώνται από πολιτικά παιχνίδια στα κράτη-μέλη. Αναφέρομαι στο κράτος δικαίου. Και γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ε, που δυνητική υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι θα ε, θεσπίσει μηχανισμό για την προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την προηγούμενη φορά δεν το τόνισε, αλλά θα ήθελα να σταθώ στην αποτυχία της Κροατίας να σεβαστεί την απόφαση του Διατητικού Δικαστηρίου. Ε, ελπίζω η επόμενη Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικεντρωθεί στο θέμα και θέλουμε να έχουμε και νομική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση του Διατητικού Δικαστηρίου. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και δεν είμαι η μόνη που επιθυμεί το σεβασμό του. Ο κύριος Ο κύριος Κρίστιαν Παρακαλώ. Υπάρχει κουμπί για το μικρόφωνο στο έδρανό σας. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Παρακαλώ, ορίστε, άνοιξε. It's on. Merci. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε για την πρώτη μου παρέμβαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ που δίνετε και το λόγο σε έναν νεοκλογιόντα, ο οποίος δεν είναι από, σαν τους υπολείπους. Είμαι Γάλλος, ε, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σκοτία στην Ευρώπη. Ήμουν βουλευτής ε, στο Κοινοβούλιο της Σκωτίας και βρίσκομαι εδώ εξαιτία του Brexit για να σας δείξω ε, πόσο συνδεδεμένοι είμαστε εμείς από την Ευρώπη. Πριν από πολλά χρόνια ψήφισα ε, το Σκοτικό Κοινοβούλιο να ε, επανέλθει μετά από μια διακοπή 30 ετών. Ένα κοινοβούλιο το οποίο ε, δεν έπαψε ποτέ, 300 ετών, δεν έπαψε ποτέ να έχει αυτό το δικαίωμα ε, μας υποστηρίξετε και δεν θα το ξεχάσουμε. Το 62% των Σκοτσέζων ψήφισαν υπέρ της παραμονής ε, της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η πιο ευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτό ε, φαίνεται στη Σκοτία γιατί έχουμε πολλαπλές ταυτότητες. Είμαι 100% Σκοτσέζος, είμαι 100% Γάλλος και 100% Ευρωπαίος. Η ιδέα μας για την Ευρώπη είναι η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, ελεύθερη ανταλλαγή κοινών αξιών και είμαστε προετοιμασμένοι να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, να μείνουμε στο επίκεντρο της Ευρώπης. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Mr. Jack Madison. Ο κύριος Τζακ Μάντισον, δεν τον βλέπω στο εδρανή του. Βρίσκεστε εδώ, στην αίθουσα, δεν νομίζω. Περνάμε λοιπόν στην κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία το Δεκέμβριο του 2015 εξέδωσε ένταλμα ψήληψης ε, ε, ε, κατά του Ράντιτα και του Βιγέριτσα Ε, με την υποψία ότι ε, προσπάθησαν να εκφοβήσουν και στη συνέχεια να εξαγοράσουν μάρτυρες. Το ε, Γενάρη του 2019 ε, εξεδόθηκε το ένταλμα. Οι αρχές του Βελιγραδίου όμως εξακολουθούν να αρνούνται την εκτέλεση της δικαστική αυτής απόφασης γιατί λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί Ε, μάλλον ε, ε, υποχρεούται να εκδώσει βάσει συμφωνία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο του εκκληματίε πολέμου, αλλά όχι εκείνου που δεν ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του. Τώρα θα πάει αυτό σε ένα διαιτητικό δικαστήριο. Μα είναι δυνατόν η Σερβία να διαμαρτύρεται κατά των ενταλμάτων σύλληψη. Για την Σερβία ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά αρνείται ανοιχτά την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χαΐς και ε, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται το άρθρο 23. Αυτό λέει πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποκρισία της. Ο κύριος Γεωργίου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έρχομαι από την Κύπρο. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του νησιού όταν η χούντα μέσα από τους σχεδιασμούς του νάτο και έχοντας τη στήριξη της ντόπια φασιστικής οργάνωσης εόκα διέπραξε πραξικόπημα αποβλέποντας τη θανάτωση του νόμιμου προέδρου αρχιεπισκόπου μακαρίου. οι συνέπειες υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι τραγικές για τον τόπο και τον λαό μας με χιλιάδες νεκρούς πολλούς μέχρι και σήμερα αγνοούμενους με μια βίαιη κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφου με έναν επικισμό και μια προσπάθεια αναλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του τόπου μα. χρειαζόμαστε και ζητούμε την έμπρακτη στήριξη τη ευρώπη μακριά από μέτρα τα οποία επαναλαμβάνονται ή αναμασούνται και είναι κατώτερα των περιστάσεων μια τουρκία η οποία φαίνεται να είναι πολύτιμη για κάποια συμφέροντα της ευρώπης όμως πολυτιμότερη είναι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου προς την κατεύθυνση να επαναρχίσουν οι συνομιλίες όπως έχουν διακοπεί από το Κράμ Μοντανά, ολοκληρώνω, για να υπάρξει μια λύση η οποία θα βοηθά τον κυπριακό λαό, τους λαούς της περιοχής, θα συμβάλει όμως και σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 400.000 ε, άνθρωποι από τα East Midlands με ε, ψήφισαν για να έρθω εδώ να τους εκπροσωπώ. 200 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη ψήφισαν για όλους εμάς ε, να μας στείλουν εδώ. Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται σε εμά, τους 751 άμεσα εκλεγμένους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούμε τους ψηφοφόρους μας εδώ στο Κοινοβούλιο όπου γίνονται οι συζητήσεις και έχει και ένα αντίστοιχο στις Βρυξέλλες. Για ποιο λόγο ε, είναι λιγότερες από 60 ημέρες ανοιχτά το ε, ημικύκλιο. Την περασμένη εβδομάδα το ημικύκλιο ήταν κλειδωμένο όλη την εβδομάδα. Σήμερα για όλο τον Ιούλιο μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα μόνο σήμερα και ορισμένοι έχουν επιλεγεί μόνο για 60 δευτερόλεπτα. Διερωτώ με, γιατί είναι τόσο λίγοι ευρωβουλευτές παρόντες, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε, μήπως ή μήπως άραγε ε, δεν θέλουν ψηφοφόροι μας να ακούγεται τη φωνή τους. Ή μήπως η πραγματική απάντηση είναι ότι ε, εκείνοι στα Συμβούλιο και στην Επιτροπή ε, πίσω από κλειστέ πόρτες δεν θέλουν να ακούσουν τι έχουμε να πούμε. 60 ημέρες δεν φτάνουν για να ακούγεται τη φωνή μας. Ούτε 60 δευτερόλεπτα φτάνουν. Οι φωνές μας θα πρέπει να ακούγονται. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα περισσότερο κοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι ότι αν όλοι υπερβαίνουν το ένα λεπτό, δεν θα καταφέρουν να μιλήσουν όλοι. Ε, σήμερα το απόγευμα δεν είναι πρόβλημα αυτό βέβαια, αλλά θα είναι πρόβλημα για το μελο... στις μελλοντικές συνεδριάσεις σας. Παρακαλώ λοιπόν μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Η κυρία Μποσκάρ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την 1η Ιουλίου στην Ουκρανία θα γίνουν πρόορες εκλογές ε, που η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Μετά τις ε, εκλογές έγιναν ε, ταχείες αλλαγές, αλλά μετά η εφραπτική ε, επιτροπή δεν έφτιαξε ουγγρική πλειοψηφία και βλέπουμε και απάτες και περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας ψηφοθυρίας και άλλου είδους καταχρήσεις. Ε, και ε, προσπάθησαν να προσελκύσουν ψήφους, ε, να δελεάσουν τους πολίτες. Ακόμη και οι μυστικές υπηρεσίες παρενοχλούν τους πολίτες που συμμετέχουν στις εκστρατείες. Δυστυχώς, οι επικεφαλής της κοινότητας στην Ουγγαρία εκτίθενται σε αυτές τις παρενοχλήσεις. Δώστε προσοχή σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή τη χώρα. Η Ουκρανία δεν πρέπει να μιλάει μόνο για την ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή, αλλά θα πρέπει να τηρεί και τα δικαιώματα και τους κανόνες. Η κυρία Κρέτσου. Εκτός μικροφώνου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω και πάλι από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να μιλήσω για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που αποτελεί την εγγύηση. Σας παρακαλώ πολύ. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι η εγγύηση μια σταθερή Ευρώπη, μια προβλέψιμη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την, τα οικονομικά και ο επόμενο προπολογισμό για το 2022-2027 δεν αντιπροσωπεύει απλά μια προτεραιότητα, αλλά είναι επίγον θέμα. Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση του προπολογισμού από το 2 Μαΐου του 2018, έγιναν μόνο τρεις διάλογοι σε αυτό το θέμα. Και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να απορούμε ότι αυξάνεται ο λαϊκισμός στην Ευρώπη. Είναι μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν έχουν διπλασιαστεί τα ποσά, εάν εγκριθούν από εσά ως συνομοθέτες και από το Συμβούλιο, για την έρευνα, για την καινοτομία, για την νεολαία, για τα προγράμματα Εράσμους, για να μην μιλήσω και για την πολιτική συνοχή που συμβάλλει στη μείωση του χάσματος ανάμεσα στις περιφέρειες και αφετέρου και για την, ε, την γεωργία. Άρα θα θέλουμε, να, θέλω να ξεκινήσουμε τον τρίλογο ε, ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το θέμα του προπολογισμού 21-27. Ε, δεν είμαι συνηθισμένη να μιλάω για ένα λεπτό, θα πρέπει να ξανασυνηθίσω. Ευχαριστώ. Όταν ε, είναι κάποιος επίτροπος έχει περισσότερο χρόνο. Λυπάμαι, ε, το κοινοβούλιο δεν δίνει τόσο πολύ χρόνο. Οι Βρετανοί συνάδελφοι θα πρέπει να λένε, ξέρουν βέβαια ότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Ε, η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα στη συνέχεια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην στο χωριό μου που είναι ε, θαλασσινή ε, χρησιμοποιούμε την έκφραση «αβάντε» και σημαίνει δύναμη, ψυχή, αλληλεγγύη. Αυτό το καταλαβαίνουν οι ε, οικογένειες ε, των ανθρώπων που επλήγησαν από φρικτές κα, και πλημμύρες στην περιοχή της Ναβάρος σε τρεις ώρες είχαμε το τριπλάσιο της βροχόπτωσης που είχαμε σε όλο το μήνα του Ιουλίου. Τρεις ε, δήμοι καταστράφηκαν ολοσχερός ε, και αυτό ε, μας κάνει να ανησυχούμε για τα ακραία ατμοσφαιρικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η ένδειξη αλληλεγγύης είναι και μία έκκληση ώστε το θέμα της κλιματικής αλλαγής να αποτελέσει προτεραιότητα σε αυτή τη θητεία. Χρειαζόμαστε μία συνολική στρατηγική σίγουρα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω, διότι πολλές από τις αποφασιστικές μάχες δίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Τσεκάρντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έναρξη αυτής της ιτίας ε, κατέστησε σαφές ότι υπάρχουν δύο αντιλήψει για την Ευρώπη. Η πρώτη είναι αυτή των γραφειοκρατών που ασχολούνται με το ευρώ, με την προστασία των ελίτ και τελικό στόχο είναι η υλοποίηση μια Ευρώπη χωρί σύνορα, χωρί ταυτότητα, η οποία θα αποτελείται από εργαζομένου ε, οι οποίοι ε, υποαμείβονται και του εκμεταλλεύονται και καταναλωτές οι οποίοι είναι έρμεο των ε, χρηματοπιστωτικών αναγκών. Η δεύτερη ε, βασίζεται στην ε, λαμπρή ιστορία αυτής της Υπήρου, η οποία βρει λόγο ύπαρξη στην προστασία των λαών μας και έχει ως τελικό στόχο την οικοδόμηση μιας Ευρώπης η οποία θα προστατεύει την ταυτότητα και τη δημοκρατία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Σασόλη που βρίσκεται στη θέση του πρόεδρου ε, γνωρίζει αυτές τις αλχημίες ε, μεταξύ ε, του ΕΛ και των σοσιαλιστών, αυτοί οι οποίοι, αυτές οι οποίες έπλεξαν και την Ιταλία και την τιμώρησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, και τιμώρησαν και τους βιοτέχνες μας, ε, του γεωργού μας και τη οικογένεια μας. Το λέω εδώ στην Ομίγυρη, αλλά κυρίως εκείνου που ακούνε εκτός ε, του Κοινοβουλίου. Δεν θα σταματήσετε την επανάστασή μας με αυτέ τι ε, συμφωνίες του Παλατιού. Η κυριαρχία του λαού θα πριτανεύσει. Ο κύριος Βόντρα βρίσκεται στην αίθουσα. Όχι. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Μποτέγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 113 εκατομμύρια Ευρωπαίων σήμερα κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια. 113 εκατομμύρια κινδυνεύουν να πέσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό δεκαπλάσιος πληθυσμός από τον πληθυσμό της χώρας μου του Βελγίου. Σήμερα υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση στα κοινωνικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση, αλλά συνέπεια των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί εδώ από τα παραδοσιακά κόμματα που μας περιστοιχίζουν, που ψήφισαν ε, απελευθέρωση, μετά την απελευθέρωση και περικοπή του προπολογισμού μετά την περικοπή του προπολογισμού. Σήμερα αυτή η λογική των ευρωπαϊκών συνθήκων που απέναντι στις ανάγκες του λαού, που απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων προσπαθεί και, και ε, προτιμά να δώσει προτεραιότητα στις αγορές είναι απαράδεκτη. Έχουμε λοιπόν την εξή επιλογή. Είτε θα συνεχίσει αυτή η κατρακύλα και εμείς θα παρακολουθούμε, είτε θα ενισχύσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις για να έχουμε μια Ευρώπη όχι της λιτότητας αλλά της ευημερίας και όχι του κοινωνικού ντάμπινγκ αλλά της κοινωνικής προόδου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Παπαδάκης παρακαλώ καταδικάζουμε τη χρησιμοποίηση δύο πλοίων με γεωτρύπανα στην κυπριακή αόζ όπως και τις διαρκείς παραβιάσεις στο αιγαίο από την αστική τάξη της τουρκίας χώρας μέλος του νάτο και στρατηγικού εταίρου της ευρωπαϊκής ένωσης που διατηρεί 45 χρόνια τώρα την κατοχή στο 37% της Κύπρου. Οι τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπλένονται με φραστικές ανησυχίες και με μέτρα που αποτελούν μέρος του γνωστού παζαριού με την αστική τάξη της Τουρκίας οι ίσες αποστάσει και τα περί από ηπα ευρωπαϊκή ένωση και νατο νομιμοποιούν την επιθετικότητα τη Τουρκία και διαμορφώνουν έδαφο για την επικίνδυνη συνδιαχείριση του αιγαίου και των κυπριακών θαλάσσιων ζωνών. η νέα κυβέρνηση τη νέα Δημοκρατία στην ελλάδα στο έδαφο που έστρωσε ο σύριζα επιταχύνει τη βαθύτερη εμπλοκή στου υπερελιστικούς σχεδιασμού, των οποίων τα μονοπόλια λιμένονται τι ενεργειακέ πηγέ κόντρα στον εφησυχασμό αλλά και τους εθνικιστικούς λεονταρισμούς οι λαοί να δυναμώσουν την επαγρύπνησή τους για την απεμπλοκή από τα υπερελιστικά σχέδια για να γίνουν κύριοι του ενεργειακού πλούτου με σχέσεις φιλίας αλληλεγγύης και κοινής πάλης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Ε, υπάρχει μια επέτειος ε, από το τέλος του Ισραηλο-Αραβικού πολέμου. Τότε οι ε, χώρες της ε, ευρωπαϊκής κοινότητας, μεταξύ αυτών ε, και η Γαλλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως ήταν η Τσεχοσλοβακία, βοήθησαν το, το Ισραήλ, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός της δημοκρατίας. Το Ισραήλ είναι από τις λίγες χώρες της περιοχής εκεί που είναι μια γνήσια δημοκρατία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις με το Ισραήλ. Γιατί ζήτησα να μιλήσω σήμερα. Διότι ανησυχώ ανησυχώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρεί στη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ και το διάλογο που έχουμε με άλλες χώρες στην περιοχή. Μα πώς είναι δυνατόν από το 2012 να μην έχει συνεδριάσει το Συμβούλιο Σύνδεσης. Αύριο θα το συζητήσω αυτό με την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βονσάλες Κασάρες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η δημόσια υγεία συνιστά τον πυρήνα και την καρδιά του κράτους δικαίου και μιας δίκαιης κοινωνίας. Για να είναι ποιοτική, χρειάζεται ανθρώπινο κεφάλαιο. Δυστυχώς, σε πολλά σημεία της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε κάποιες περιφέρειες της Ισπανίας, ε, στην Γαλλικία έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και άλλα επαγγέλματα υγειονομικά. Ε, γίνονται πραγματικά ε, μεγάλες καταχρήσεις από τη Σούντα Ντεγαλίσια που είναι η ντόπια κυβέρνηση. Ε, οργανώνονται οι νοσηλεύτριες ε, για ε, να αντισταθούν στον αγώνα Τη κυβέρνηση εναντίον του. Μέχρι και 500 συμβάσεις έχει υπογράψει νοσοκόμα μέσα σε μία δεκαετία. Γι' αυτό στην παρθενική μου ομιλία εδώ θέλω να τονίσω ε, ε, τη σημασία του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που απαιτούν σεβασμό, αξιοπρέπεια και σωστές συνθήκες ε, για να ασκήσουν το επάγγελμά του. Ευχαριστώ. Mr. Flago. Για μένα η Ευρώπη είχε πάντα και ε, πρέπει να εξακολουθήσει να έχει ένα ε, ισχυρό πνεύμα ανοχής και προοδευτικότητας. Δυστυχώς σήμερα ε, με τις τεχνολογικές πρόοδους και τα επιτέγματα που χρειάζονται για τον έλεγχο των συνόρων η Σλοβενία και η Ιταλία, οι γείτονέ μας, έχουν ανακοινώσει νέα χιλιόμετρα σειρματοπλέγματος στα σύνορά μας. Είμαστε ε, εναντίον αυτού, διότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Ε, αυτό σημαίνει περισσότερους πολέμους, περισσότερα συμμερτοπλέγματα και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι εντελώς λαθασμένη προσέγγιση. Θα πρέπει φυσικά να ε, προσέξουμε το θέμα της ασφάλειας. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε ε, για το θέμα των μεταναστών και να τους μεταχειριζόμαστε με ανθρωπιστικό τρόπο. Αλλά τα συμμερτοπλέγματα δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Κομισιόν είναι να βρει έναν τρόπο να πολεμήσει την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Θα πρέπει να το λύσουμε σύντομα αυτό. Ο κύριος Φέστ. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ συζητάτε για την υψηλή πολιτική. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η συμπεριφορά του Κοινοβουλίου εδώ. Ε, καταρχήν, οι βουλευτές ε, ορίζουν την πολιτική ατζέντα και το πρόγραμμα. Οι βουλευτές αποφασίζουν τα πολιτικά θέματα και τις πρωτοβουλίες με τις οποίες θέλουν να ασχοληθούν. Αυτό δυστυχώς παραβιάζεται. Σήμερα πήρα ένα έγγραφο, ο κύριος Κλάους Βέλε μάλλον είναι ο υπεύθυνος της σύνταξης που είναι η διοίκηση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Εσωτερικών Υποθέσεων και Ελευθεριών και φέρει τον τίτλο «Πιθανές πρώτες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες» και ασχολείται με διάφορα θέματα ε, για τα οποία μας έχουν στείλει εδώ οι πολίτες να τα αποτρέψουμε. Ε, με την κατάσταση, επανεκατάσταση, ανθρωπιστικές θεωρήσεις, ε, ΜΚΟ κτλ. Φαίνεται να πιστεύει η διοίκηση ότι το πολιτικό θεματολόγιο και το πρόγραμμα δεν το ορίζουν οι βουλευτές, αλλά η διοίκηση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ασέβεια και σας παρακαλώ να ψάξετε πόσα χρήματα έχουν αφιερώσει σε αυτό το πράγμα και πώς μπορούμε στο μέλλον να τα αποφύγουμε και να τα αποτρέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, ξέρετε, είμαι μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας και θα ήθελα να εκφράσω μια πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία που έχω ε, ε, σχετικά με την εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Τώρα, δεν θα πρέπει βία να επιβάλλουμε αυτή τη συμφωνία επειδή έχει τραβήξει μια 20 αυτή η υπόθεση και θα πρέπει να τελειώνει. Στη Γαλλία και στην Πολωνία και τα λοιπά ε, είναι πολύ σημαντική η αγορά ε, και θα διαταραχθεί η αγορά γεωργικών προϊόντων, κρέατος όπως είναι το χείριο κρέας κτλ. που έτσι κι αλλιώς θα κλονιστεί λόγω και του Brexit. Ε, δεν έχουμε ε, τις ίδιες προδιαγραφές με τις χώρες μερκοσουρ, ούτε υγειονομικές, ούτε περιβαλλοντικές και το πρόβλημα το έχουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Ελπίζω να μην εφαρμοστεί η συμφωνία πριν κυρωθεί και πριν τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγες μέρες μετά τις ε, εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις συστάσεις αναχώρα οι οποίε προβλέπουν κυρώσει για τα κράτη-μέλη, για να είμαστε κατανοητοί περί τίνο πρόκειται. Δεν υπάρχουν μεγάλε αλλαγέ ε, εκτό από κάτι καινούριο για την Πορτοκαλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει περισσότερο ε, περικοπέ ε, στον προπολογισμό. Επομένω, θέλουμε να μειώσουμε τι μεταφορέ, τον πολιτισμό, την παιδεία, τη στέγαση και οι πόροι αυτοί φυσικά θα τους στερηθούν οι εργαζόμενοι της Πορτογαλίας και θα τους πάρουν αυτοί οι οποίοι κερδοσκόπησαν πάνω στην υποτίμηση της χώρας. Ε, μεγαλύτερη επισφάλεια. Αυτό σημαίνει το να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας και να μειώσουμε και προς τα κάτω τις συνθήκες εργασίας. Ε, σήμερα, αυτές τις μέρες συζητείται πολύ ποιος ε, θα αναλάβει ε, τα καθήκοντα και τα πόστα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έχει σημασία είναι να αλλάξει η πολιτική. Δεν έχει σημασία ποιος κρατάει τα σκύπτρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις πολιτικές, γιατί τις πολιτικές πρέπει να αλλάξουμε. Επόμενος ομιλητής, κυρία Βριονίτη Βόζεμπεργκ. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην περασμένη θητεία απασχόλησε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το πολύ σημαντικό θέμα της μετανάστευσης είμαι από την ελλάδα και ξέρετε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα. η νέα κυβέρνηση της ελλάδος εγγυάται την αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για μια υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική. όμως έχουμε μπροστά μας δύο προβλήματα. το ένα αφορά στην μη αναθεώρηση του κανονισμού του δουβλίνου που έχει μείνει στο συμβούλιο και το δεύτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα αφορά σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν κλείσει τις πόρτες τους και δεν δέχονται να εφαρμόσουν τις κοινέ μας αποφάσεις δεν δέχονται την ανάληψη κοινών ευθυνών δεν βοηθούν ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα αντιμετώπισης του ασύλου έτσι ώστε να μην κλονίζεται η αξιοπιστία των ευρωπαίων πολιτών και να μην συνηγορούμε στο να ρίχνουμε λάδι στο μήλο του λαϊκισμού. σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία μου. Ε, κυρία Βόλτερ, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το περασμένο μήνα ε, μου άρεσε ε, πολύ ε, η ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου, εθνική ομάδα της Ολλανδίας οι ε, πορτοκαλί λένες. Μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστο αυτό το άθλημα και άγνωστη και η ομάδα. Όπω ήταν άγνωστοι και οι ευρωεκλογέ. Όμω η κλιματική αλλαγή, το Brexit και η άνοδο ε, του εθνικισμού αφύπνισε του λαού και τον κόσμο. Και είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή εδώ και δεκαετίε στι ευρωεκλογέ και ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι νέοι δεν ψήφισαν την Ούρσο Φόντερ Λάιν, ψήφισαν υποψηφίους που πριν τις εκλογές ξεκαθάρισαν τη θέση τους και άνοιξαν τα χαρτιά τους. Φανταστείτε ο τελικός ε, του παγκοσμίου κυπέλου ε, ποδοσφαίρου, ε, του παγκοσμίου πρωταθλήματος που ήταν αντίπαλες ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και κάτω χωρών, έχει κερδιθεί από τη Γαλλία, που δεν συμμετείχε ε, καν στον τελικό. Εγώ δεν θα ψηφίσω την κυρία Φόντερ Λάιεν, ούτε την υποψήφια της Καμαρίλας, γιατί δεν είναι αυτή η υποψήφια που θα πρέπει να εκλέγονται πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κόφουντ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλησα να πάρω σήμερα το λόγο, διότι ε, χάσαμε την περασμένη εβδομάδα μια υπόθεση στο δικαστήριο των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τορπίλησε τη στεναρή πολιτική σε θέματα μετανάστευσης. Μα αυτό είναι γελίο. Ε, οι Δανείοι ποτέ ε, δεν δέχτηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί στα εσωτερικά της θέματα. Εδώ ε, και τα τελευταία χρόνια στο Folketing στη Βουλή μας έχουμε πλειοψηφία ε, για μια ε, στεναρή πολιτική στη μετανάστευση. Ξέρετε, η Δανία ανήκει στους Δανούς ε, θα πρέπει κάποιο να πληρεί κάποια κριτήρια για να έρχεται στη Δανία. Είναι πραγματικά χονδροειδή ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαστηρίου ε, και ε, στρέφεται κατά της αυτοδιάθεσης του δανικού λαού. Ο κύριο Μπούντα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Οι Ρουμάνοι αγρότες χρειάζονται σταθερή και ταχεία απάντηση σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που διαπραγματεύομαστε την σύσταση της Νέας Επιτροπής, ζητώ δημόσια από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μην χρησιμοποιούν τον κανονισμό για την ΠΑΚ ως αντάλλαγμα για να πετύχουν άλλους πολιτικούς στόχους. Ε, ε, το την προσοχή όλων των ηθήνοντων των πολιτικών να μην παίζουν με τις μοίρες των αγροτών, των Ρουμάνων και Ευρωπαίων αγροτών που χρειάζονται σταθερότητα. Αυτός ο κανονισμός ε, είναι σημαντικός, αντιστοιχεί σε σημαντικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των μεγάλων και μικρών αγροτών και είναι και θετικό και για τους καταναλωτές για να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα ποιότητας και λογικές τομές, τιμές. Ε, άρα η μόνη λύση είναι να αποσταλεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής του, του Ευρωκοινοβουλίου. Τα κράτη-μέρη θα πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο για να υιοθετήσουν τα στρατηγικά εθνικά τους σχέδια. Ευχαριστώ. Η κυρία Κυρία Πρόεδρε, Παρά το γεγονό ότι είμαστε διαρριμμένοι ω Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία είναι ζωτική σημασία για την καταπολέμηση τη σύγχρονη δουλεία. Η διακίνηση ανθρώπων, η καταναγκαστική εργασία ε, και τα σεξουαλικά εγκλήματα αφορούν εκατομμύρια ανθρώπου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο ρυθμό καταγεγραμμένων θυμάτων και η βορειοανατολική πλευρά έχει το υψηλότερο ποσοστό προβλήματο εκτό του Λονδίνου. Ταυτόχρονα όμω είμαστε και παγκόσμιο ηγέτη ε, στην ομοθεσία για τη σύγχρονη δουλεία και τη δράση. Γι' αυτό έχει σημασία ε, ε, ο επόμενος, ε, το γεγονός ότι ο επόμενος επίτροπος κατά του εγκλήματος στην Ορθούμπρια έχει προχωρήσει τα θέματα αυτά. πρέπει να συνεργαζόμαστε περιφερειακά και ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εκριζώσουμε αυτό τη μορφή εγκλήματος που δεν ανήκει στο σύγχρονο κόσμο και θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε το Brexit να μας κατρακυλήσει σε αυτό το παρελθόν. Ευχαριστώ κύριος Μπόγκοβιτς. Η Σλοβενία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες ε, με την αύξηση των επιθώσεων από λύκους και αρκούδες ε, κατά κατοικίδιων ε, και οικόσιτων ζώων. Έχουμε πάνω από 100 πρόβατα τα οποία σφαγιάστηκαν, ε, το ίδιο και αγελάδες, ακόμα και επίθεση σε μια γυναίκα είχαμε. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση στον αριθμό αυτών των άγριων ζώων και τα τελευταία χρόνια γεννιούνται περισσότερα ζώα από όσα θανατώνονται. Οι αγρότες χάνουν την ελπίδα τους ε, και οι κτηνοτρόφοι πλέον ε, λένε ότι η μόνη λύση είναι να εγκαταλείψουν αυτή τη δραστηριότητα. Το Υπουργείο Γεωργίας λοιπόν στη Σλοβενία πρότεινε νομοθεσία για εξαιρετικά μέτρα κυνηγιού για ε, λύκους και αρκούδες. Θεωρώ ότι το θέμα όμως θα πρέπει να συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πλήξει μόνο τη Σλοβενία, ε, πλήττει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι συνέπεια της διαταραχής της ισορροπίας της φύσης. Και επομένως, ε, ε, επειδή έχει συμβεί στη Σλοβενία, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί θα συμβεί και σε όλες τις χώρες. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να εξαπλωθεί το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλα μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο, αλλά δεν έχουν έλθει ακόμα στην αίθουσα. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν ο... η σύνοδος του ενός λεπτού. Ε... Διακόπτεται η συνεδρίαση. Απλώ να πω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι αύριο, ε, Τρίτη, 9 η ώρα. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα. Καλό σας βράδυ.